πριν να γκρεμίσουμε τους τοίχου που χώριζαν την Ευρώπη, πριν δημιουργήσουμε μια οικονομική και νομισματική ένωση και πριν ανοίξουμε τα σύνορα, μεγαλώσαμε με μια τεράστια πολιτιστική, κινηματογραφική κληρονομιά, μια κληρονομιά κοινή που μας ενώνει όλους, που μας κάνει όλους πιο Ευρωπαίους. Είμαστε το μόνο κοινοβούλιο στον κόσμο που απονέμει ένα κινηματογραφικό βραβείο. Και οι τρεις ταινίε ε, που είχατε την ευκαιρία να δείτε αυτές τις τελευταίες εβδομάδες υποτιτλίστηκαν σε 24 γλώσσες και προβλήθηκαν και στις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, προβολές και συζητήσεις ε, πολλές φορές ταυτόχρονα οργανώθηκαν σε 46 διαφορετικές πόλεις και μαζί με το πρόγραμμα Creative Europe της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ήθελα να ευχαριστήσω ειλικρινά όλους όσοι πρόθεσαν ε, και ανέπτυξαν και έδωσαν τη δυνατότητα στους ε, σκηνοθέτες μας, στους κινηματογραφιστές μας να ε, συνδιαλλαγούν με τους λαούς μας. Θα ήθελα να αποτύσω φοροτιμή στο θάρρος των σκηνοθετών που βρίσκονται εδώ σήμερα. Όταν καταφέρνουμε να πάμε στον κινηματογράφο, αντιλαμβανόμαστε, βλέπουμε το τελικό προϊόν. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλα αυτά είναι το αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, πάθους, ε, πολλών προσπαθειών και μερικές φορές και κινδύνων. Κινδύνων που διατρέχουν πάρα πολλοί ε, σκηνοθέτες ε, και παραγωγή στη δουλειά τους. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και το θάρρος αντιμετώπισης ζητημάτων μερικές φορές δύσκολων πολιτικής επικαιρότητα. Μην ξεχνάμε την, το διαρκή αγώνα για την ελευθερία της έκφρασης και τη δημιουργικότητα. Υπενθυμίζω σε όλου ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δεσμευτεί στη συζήτηση για το copyright να υπερασπίζεται τα δικαιώματα του δημιουργού. Και φυσικά καλό και τα εθνικά κοινοβούλια να την κυρώσουν το συντομότερο δυνατόν. Οι σκηνοθέτε, οι κινηματογραφιστέ που είχαμε την τιμή να γνωρίσουμε στο πλαίσιο του βραβείου Λουξ ε, μα κάνουν περήφανου. Ζήτω λοιπόν η ελευθερία έκφρασης. Ζήτω ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος Ζήτω οι κινηματογραφιστές μα οι σκηνοθέτε μα που βρίσκονται εδώ σήμερα μαζί μα. Ευχαριστώ. Αυτός είναι ο φάκελο. Allora. God exists. Ο Θεός υπάρχει. Το όνομά της είναι Πετρούνια. Η κυρία Τεώνα Στρούγκαρ Μητεύσκα. Actually, I prepared something. I ask you for your patience. Sorry, it's a very exciting moment. Είναι μια εξαίρετη στιγμή για μένα. Πετρούνια. Η πετρούνια είναι μία θα έλεγα τολμηρή, ζωηρή, γενναία, παλεύει για τη δικαιοσύνη, δίνει αγώνα για τη δικαιοσύνη και ο αγώνας αυτός μας ε, κάνει να συγκινηθούμε. Πάντα μου λένε οι πολιτικοί στη χώρα μου ότι τα έργα μου είναι ιδιαίτερα πολιτικά. Εμένα με ενδιαφέρουν όμως τα κοινωνικά φαινόμενα και γι' αυτό θέλω να λέω τη γνώμη μου και να μιλάω για προβλήματα τα οποία πολλοί δεν θέλουν να θέσουν. Γιατί πώς ε, θα μιλήσουμε για το μέλλον της χώρας μας αν δεν μιλήσουμε για τα προβλήματα. Θα πρέπει λοιπόν να εκφράζουμε ελεύθερα τις απόψεις μας και γι' αυτό ζητώ από εσά τους πολιτικούς εξ ονόματος όλων των παραγωγών, σκηνοθετών και συντελεστών στον κινηματογράφο να διασφαλίσουν τα δικαιώματά μας, την ελευθερία έκφρασης και την ελευθερία του λόγου από τη στιγμή που έφτεσα εδώ χθε, ε, γνώρισα ιστορίες, άκουσα ιστορίες για ανθρώπους που πέρασαν ε, χρόνια στη φυλακή ε, για λόγους παραβίασης των ελευθεριών τους. Αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει. Πρέπει να κρατήσουμε λοιπόν, να έχουμε την ελευθερία έκφρασης χωρίς κανένα φόβο. Είμαι γυναίκα, είμαι από τη Βόρεια Μακεδονία και είμαι Ευρωπαία και πιστεύω στο μέλλον της Ευρώπης ε, στα πλαίσια της αλληλεγγύης και της συμπερίληψης και όχι του αποκλεισμού. Είμαι γυναίκα, είμαι από τη Βόρεια Μακεδονία, είμαι Ευρωπαία και το μέλλον της Ευρώπης βρίσκεται στην αλληλεγγύη και στη συμπερίληψη και όχι στον αποκλεισμό. Σας ευχαριστώ. Να συνεχίσουμε, γιατί σήμερα υπάρχουν και άλλοι νικητές. Θα δώσουμε την ευκαιρία και στους άλλους ε, φυσικά και συγχαίρω και εγώ την ε, Πετρούνια και χαίρομαι πάρα πολύ. Τρει όμω είναι οι σημερινοί νικητέ. Οπότε ο δεύτερο νικητή ή ο εξίσου νικητή σήμερα είναι. Cold case Hammersholt. Cold case Hammersholt. Κλειστό φάκελο Hammersholt. Συγχαρητήρια. Και μην φύγετε ακόμα γιατί υπάρχει και ένα τρίτο βραβείο. Και ο τρίτος ε, νικητής, μια πάρα πολύ όμορφη ταινία και ξέρω ότι έγιναν πάρα πολλές συζητήσεις και εδώ ε, στο σώμα αυτό. Το τρίτο βραβείο λοιπόν πηγαίνει, εντάξει ξέρουμε σε ποιον, στην ταινία El Reino, έκπτωτος. Παρακαλώ. Ο Ροντρίγκο.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 Γεια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 πίσω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

Ο κύριος Γκέι καταλάβει. Τα Ah,